για τις ε, Ολομέλειες του 2017 στην ε, συνεδρίαση της η διάσκεψη των Προέδρων υιοθέτησε το σχέδιο προγράμματος είναι διαθέσιμες οι συνεδριάσεις στις ιστοσελίδες η προθεσμία για πρωτοβουλίες είναι 3η 6 Οκτωβρίου στις 12 ε, το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 12.30 η πρόεδρος έλαβε από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές έτοιμα άρσης ασυλίας για τον κύριο Σικέρσκι